Αγαπητοί συνάδελφοι. Α. Äh, Σας ε, καλωσορίζω στη σημερινή μας συνεδρίαση όπου θέλουμε να ψηφίσουμε την τελική έκθεση της Περβών Περές αλλά προτού προχωρήσουμε ή στη ψηφοφορία θέλω να, κάνουμε θέλω να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις και να δώσω σύντομα το λόγο και στην Περβών διότι αυτό το οποίο πετύχαμε σήμερα δηλαδή να φτάσουμε στην ψηφοφορία της έκθεσης ε, είναι ε, κάτι το οποίο οφείλουμε σε διάφορους συνεργάτες Επιτροπής μας, ιδίως της ε, Περμός αλλά και των συντονιστών και της Γραμματείας. Ε, διότι θέλω εδώ να την επενέσω, έκανε ό,τι ήταν δυνατόν και αναγκαίο. Βεβαίως, κοιτάζοντας τα κείμενα το τελευταίο εξαμήνου, βλέπουμε ότι έχουμε έναν πλούτο εγγράφων και πριν από το τέλος του καλοκαιριού πρέπει να υπάρξει μία τεκμηρίωση των εργασιών μας μορφή βιβλίου. Πρέπει δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του εγγράφου αυτού μέχρι τέλος Ιουλίου. Τα briefing notes, οι σημειώσεις όλα θα συγκεντρωθούν κατά τρόπον ώστε όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να διαβάζει το έγγραφο αυτό. Θέλουμε εδώ να έχουμε και τις φωτογραφίες των μελών της επιστροφής, γι' αυτό και στο τέλος θα σας παρακαλούσα να μείνετε ένα δεκάλεπτο, διότι έχουμε ζητήσει από το φωτογράφο του Κοινοβουλίου να έρθει εδώ και θα παρακαλούσα τα μέλη της Επιτροπής, όχι τους επισκέπτες, αλλά τα μέλη να παραμείνουν για να βγάλουμε μία φωτογραφία. Και τέλος, πριν από την ψηφοφορία στην Ολομέλεια, Τη της εκθέσεως αυτής. Λίγο πιο σιγά παρακαλώ, ησυχία. Θέλουμε η δουλειά μας να στεφθεί με μία μικρή δεξίωση στο Στρασβούργο με κάποια ποτά και σνακ. Αυτό θα γίνει την Τετάρτη της εβδομάδος του Στρασβούργου του Ιουλίου και την Τρίτη θα γίνει η συζήτηση της εκθέσεως στην Ολομέλεια και την Πέμπτη η ψηφοφορία. Αλλά δεν μπορώ να σας δώσω τελικές λεπτομέρειες, θα σας κοινοποιηθούν εν καιρό. Κατόπιν αυτού παρακαλώ την Περβόνς να μας πει με λίγα λόγια τη θέση της. Σε ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων που συνόδευσαν την εργασία αυτή για 18 ολόκληρους μήνες για την επεξεργασία της δεύτερης αυτής έκθεσης. Νομίζω ότι οι προτάσεις που κάνουμε είναι δυνατές προτάσεις, αυτές που κάναμε στην πρώτη έκθεση είναι δυνατές προτάσεις και κάτι μου λέει ότι και σήμερα πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και θα προχωρήσουμε με εξίσου αποφασιστικές προτάσεις. Δεν θα γίνει τώρα συζήτηση για την ουσία της υπόθεσης, αλλά θα προετοιμάσουμε λίγο την ψηφοφορία και γι' αυτό θα ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις εδώ. Πρώτον, θα ήθελα να ζητήσω η Γραμματεία να μην μοιράσει το κείμενο επί τη βάση της ψηφοφορίας που θα γίνει σήμερα, γιατί το κείμενο αυτό έχει ανάγκη, θα έλεγα, τακτοποίησης, καθαρίσματος σε εισαγωγικά και γι' αυτό πριν από το τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να γίνει μία συνάντηση η οποία να επιτρέψει να διαγράψουμε τις επικαλύψεις, τις επαναλήψεις, να βελτιώσουμε τις διατυπώσεις χωρίς φυσικά σε καμία περίπτωση να θίξουμε το νόημα και να αλλάξουμε επίσης και τη σειρά ορισμένων παραγράφων που απαιτεί το σύνολο της παρουσίας των υπαλλήλων των πολιτικών ομάδων. Θα έχει δουλειά. Γι' αυτό ζητώ συγγνώμη, αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό θα είχαμε ένα κείμενο διόλου εύπεπτο. Τώρα, μέχρι την παράγραφο 38, ο κατάλογος ψηφοφορίας δεν προσαρμόζεται απόλυτα στην πραγματικότητα που έχουμε μπροστά μας. Τι εννοώ, στην παράγραφο 17 Αν πάρετε τη συμβιβαστική πρόταση, η οποία σας έχει ήδη διανεμηθεί, Θα πρέπει να ψηφίσουμε επαναλαμβάνει η κυρία Μπερές, θα πρέπει να ψηφίσουμε τις παραγράφους δε, στο κείμενο που έχετε μπροστά σας, 17 δε λατινικό και α και την παράγραφο 17 ολόκληρη. Αυτό τι σημαίνει. Ζητώ συγγνώμη, λέει η κυρία Μπερές, έχει υπάρχει μια μικρή σύγχυση, σταμάτησε την ε, παρουσίασή της. Ce qui signifie que le... Euh, λοιπόν, τα ξαναλέμε. Το 18β δεν υπάρχει σε κανέναν από τους καταλόγους ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια ειδική ψηφοφορία για το 17β. Για, τις παραγράφους, για την παράγραφο μάλλον 48α. Θα πρέπει επίσης να πάρουμε μία απόφαση για την 48 Β. Επαναλαμβάνω ότι η 421 έχει παρουσιαστεί σαν μία παράγραφο 48 β μικρό. είναι η παλιά τροπολογία 421 και δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους ψηφοφορίας που έχετε μπροστά σας. Εκεί περιλαμβάνεται η 48α και λέγεται ότι αν γίνει δεκτή, γίνεται δεκτή και η 421. Λοιπόν, ε, ε, δεν τελείωσα πρόεδρε. Τώρα πάνω στον κατάλογο των ψηφοφοριών έτσι όπως έχει ε, διανεμηθεί στους συναδέλφους. Έγινε σε συμφωνία με τους συντονιστές, προσθέθηκαν ορισμένες τροπολογίες που θα ψηφιστούν ξεχωριστά. Κάποιες από τις τροπολογίες αυτές καλύπτονται πλήρως, οπότε δεν θα πρέπει να τις θέσουμε σε ψηφοφορία εφόσον γίνουν δεκτές οι συμβιβαστικές. Ενώ την 426, η οποία περιλαμβάνεται στο 29D αγγλικό. Δέλτα αν θέλετε, 29 Δέλτα για την 426. Ah oui, non, ça c'est η 227 του Πασκάλ Κομφά καλύπτεται πλήρως από την 27 Β μικρό νέο. Πρόκειται για την 313 του Γκαρσία Μαργάιο που καλύπτεται από την παράγραφο 27 Γ νέο. Επίσης η 421 του Κοφεράτη η οποία καλύπτεται από την 48. 48 Β, παράγραφο 48 Β, εννοώ λέει η κυρία Μπερές, η 14 του Πασκάλ Κομφά, η οποία κατά το πρώτο της τμήμα καλύπτεται από την παράγραφο D, A, νέο, αγγλικά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Αυτές ήταν οι μόνες σημαντικές παρατηρήσεις. Ίσως να υπάρχει μια τελευταία παρατήρηση εδώ, η οποία αφορά λίγο την ουσία. Σχετικά με την συμβιβαστική πρόταση για τις παραγράφους 20 και 21. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ότμα Κάρας για την εντατική του συνεργασία που μας επέτρεψε να βελτιώσουμε τη διατύπωση του κειμένου και να έχουμε ένα κείμενο που, αρμόζει, που ταιριάζει σε όλους. Χάσαμε όμως μία αναφορά στην ομάδα των 20. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας προτείνω η νέα παράγραφος 20 να αναγνωστεί με τον εξής τρόπο. θα διαβάσω μόνο το ενδιάμεσο κομμάτι, που είναι το κομμάτι επί του οποίου υπήρξε η συμβιβαστική πρόταση που έχετε μπροστά σας σήμερα. Ζητάμε την περαιτέρω ολοκλήρωση των θεσμών του Bretton Woods και της μιας δομής παγκόσμιας διακυβέρνησης οικονομικής που να περιλαμβάνει την ομάδα των 20 στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Δηλαδή ουσιαστικά ζητάνε να περιληφθεί η ομάδα των 20 στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών. Colleagues, uh, let me just, uh, uh, Συνάδελφοι, Σαν πρόεδρος της συνεδριάσεως θα πρέπει να, να σχολιάσω αυτά που είπε η Περβόνς. Καταρχήν, όπως είπε η Περβόνς, οι γλωσσικές αλλαγές πρέπει να γίνουν κατά τρόπον ώστε και η ε, ε, η διατύπωση να είναι σωστή. Αλλά θα πρέπει οι αλλαγές αυτές να ε, περιοριστούν στο γλωσσικό τμήμα. Δηλαδή ε, ε, κάποιο το, κάποιος αγγλόφωνος να θεωρεί ότι οι αλλαγές αυτές είναι απαραίτητες. Δηλαδή δεν θέλουμε να αλλάξουμε ούτε τα συμφραζόμενα ούτε το νόημα του κειμένου. Δεύτερο, όσον αφορά το 17β θα ψηφιστεί διότι δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. Η μόνη λοιπόν ερώτηση, μάλλον υπάρχουν δύο ερωτήσεις οι, περίπου οι 30 τροπολογίες εκ των οποίων ε, οι συντάκτες ζήτησαν να ψηφιστούν χωριστά στο τέλος ε, της συνεδριάσεως, στο τέλος του καταλόγου και η λέγει ότι πολλά από αυτά τα θέματα έχουν επιληθεί ε, κατά κάποιον τρόπο με τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Δεν έχω όμως πρόβλημα να τις θέσω προς ψηφοφορία διότι εφόσον έχουμε συμφωνήσει με τους συντονιστές και τις πολιτικές ομάδες. Εγώ από ό,τι ερμηνεύω περβώς πιστεύω ότι θα απορριφθούν. Δεν μας δημιουργούν όμως πρόβλημα. Άρα το μόνο το οποίο παραμένει είναι το ερώτημα εάν θα υπάρξει αναμόρφωση της προτάσεως που αναφερόμαστε στο G20 και αν θα αποτελέσουν μέρος της ευρείας μονάδας διακυβέρνησης διότι αυτό το οποίο έχουμε μπροστά μας είναι ε, σαν κείμενο είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς ε, ε, συζητήσεων μεταξύ συντονιστών, σκιωδών εισηγητών, πολλαπλών συζητήσεων. Εξώ, εξού και θα ήθελα να ψηφίσουμε. Ποιος θέλει να ψηφίσουμε βάσει του ότι έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι αυτή είναι η πλειοψηφία. Κύριε Πρόεδρε, Αντιλαμβάνουμε ότι όλοι έχουν κινητοποιηθεί για αυτή την ψηφοφορία και έχουν και άλλα να κάνουν. Αλλά ολοκληρώνουμε τις εργασίες μιας επιτροπής που αναφέρεται στην κρίση και το G20 εις ε, την ε, έκβαση των συζητήσεων αυτό για την κρίση είναι σημαντικό. Είπατε ότι πολλά από αυτά τα θέματα έχουν διαπραγματευτεί πολύ σύντομα και μόλις ε, είπα στον ε, Ότμα Κάρας ε, μία προφορική τροπολογία η οποία δεν τον προβληματίζει εάν δεν περιλάβουμε λοιπόν αυτή την προφορική τροπολογία θα παραπέμπουμε σε μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς να αναφερόμαστε στο G20. Ε, Ότμαρ, στην τροπολογία 20 δεν μπορούμε να αναφερθούμε ρητός στους G20, στο Corrigendum, στη διόρθωση, στη New Version, στη νέα μορφή της, στην πρόταση της τροπολογίας. Εγώ θα ακολουθούσα αυτή την πρόταση. Εντάξει. Συνάδελφοι, όλα έχει το λόγο. Η αναφορά στο G20 παραμένει ή όχι. Δεν το βλέπω στο κείμενο αυτό. Θα ήθελα να ξέρω εάν αφαιρείται ή όχι. Ε, παρακαλώ θα ξαναδιαβαστεί. Ε, καλεί ε, την ε, αναβίωση του θεσμού του Bretton Woods και την ένταξη του G20 στο νέο σύστημα. Και στο τέλος, στο τέλος της, του καταλόγου ψηφοφορίας έχετε την νέα συμβιβαστική πρόταση για την παράγραφο 20 ε, αλλά στη σελίδα 14 του καταλόγου ψηφοφοριών αλλά δεν αναφέρεται στο G20 ε, μιλάμε ε, για την παράγραφο 20 των διορθώσεων το, το κείμενο που λέει Corrigendum 35 του 2011 Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κάρας εδώ δεν θέλω να ενισχύσω το χάος και να δημιουργήσω σύγχυση, αλλά ε, όλα αυτά τα συζητήσαμε εν ηρεμία την περασμένη εβδομάδα. Προβλέψαμε μία ημερομηνία για την... Ε, ε, ε, ε, για τα διάφορα θέματα το, η γραμματεία τα ενσωμάτωσε και υπήρξαν διευκρινήσεις και τα δύο, σε δύο ακόμη σημεία δηλαδή ε, εάν λείπει κάτι κατά τη γνώμη της ε, ε, εισηγητρίας από το κείμενο αυτό μπορούμε όλοι μαζί να το παρουσιάσουμε στην Ολομέλεια. Αλλά εδώ μιλήσαμε ότι θέλαμε να μιλάμε για την Global Economic Governance αντί για το το G20 το προωθήσαμε την έκφραση G20 ως Global Economic Governance και αυτή ήταν η ουσιαστική σκέψη την οποία είχαμε στο μυαλό μας και συζητήσαμε δηλαδή η περαιτέρω εξέλιξη του G20 να γίνει ένα όργανο παγκοσμίου οικονομικής διακυβέρνησης ε, στα πλαίσια του ΟΗΕ. Ε, αν λοιπόν υπάρχει μία διατύπωση διαφορετική ε, μπορούμε να την περιλάβουμε στην Ολομέλεια χωρίς να αλλάζει πρόταση. Ε, επίσης το 17β ε, δεν περιλαμβάνεται εδώ και θα πρέπει να ψηφιστεί ο μπλοκ αλλά όλα τα υπόλοιπα περιλαμβάνονται και είναι εντάξει. Λοιπόν, Τώρα νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Θα κάνουμε καταρχήν μία δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε εάν ε, οι διάφορες ομάδες ε, ε, μπορούν να προχωρήσουν. Ποιος δεν έχει την κάρτα του μαζί. Λοιπόν, προτείνω να ψηφίσουμε ως των διανατάσεως χειρών. Όταν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα θα ψηφίσουμε με την κάρτα και στο τέλος θα ψηφίσουμε όχι για ονομαστική ψηφοφορία με την κάρτα αλλά απλούστατα ε, για να υπάρχει ε, η καταμέτρηση. Λοιπόν, το 17 θα συμπληρωθεί, θα ψηφιστεί επιπλέον και η παράγραφος 20. Ποιος είναι υπέρ. Ε, αντίθετη αποχές, μία αποχή βλέπω. Εντάξει. Τώρα ερχόμαστε στην συμβιβαστική τροπολογία παράγραφος 4. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Ε, συμβιβαστική παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 9β νέων. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική παράγραφος 13, πρώτο τμήμα με χωριστή ψηφοφορία που έχει ζητήσει η ομάδα των φιλελευθέρων, πρώτο μέρος, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, το υπόλοιπο κείμενο, υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Ερχόμαστε τώρα στην ε, νέα συμβιβαστική παράγραφο 17α που αποτελείται από διάφορα τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα. Η λέξη free, ελεύθερος, υπέρ. Κατά αποχές. Θα ήθελα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά γιατί είναι, δεν είναι σαφές. Λίγη ψηφοφορία. 24 επί ε, υπέρ 16 κατά εγκρίνεται. Τέταρτο μέλος, η τελευταία φράση call for the dismantling of the trade barriers. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Άποχες. Και πάλι να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο γιατί μου φαίνεται πολύ τσιματσίμα. 25 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Τελευταίο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην παράγραφο 19. Πρώτο τμήμα. Μέχρι, χωρίς τη λέξη free, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα με τη λέξη free, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στην παράγραφο 21. Έχουμε και πάλι μία διόρθωση η οποία θα ψηφιστεί καταρχήν η οποία είναι ίδια με το τέταρτο μέρος στον κατάλογο ψηφοφορία, δηλαδή ε, calls for the G20 countries του promptly adopt global coordinated policy action in order to contribute to the strong table είναι η παράγραφος 21. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 27C. Και πάλι χωριστή ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα. ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ήθελα να κάνουμε ένα ηλεκτρονικό έλεγχο. Οι 24 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Το 29D πάλι σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. η τροπολογία 34 ε, εδάφιο 4 υπέρ κατά εγκρίνεται ε, το 4C νέων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική παράγραφος 37 2α νέων και πάλι σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα χωρίς τα τμήματα 2 και 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα είναι η λέξη great υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο ε, ε, συμβιβαστική παράγραφο 37α νέων υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική παράγραφος 38 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. απορρίφθηκε 16 υπέρ 21 κατά. Συμβιβαστική 41 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε. Είναι ασαφές. Απερίφθη. 16 υπέρ, 26 κατά. Τώρα έρχομαι στην εναλλακτική ε, πρόταση του ΕΛΚ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Με συγχωρείς, Περμός, έχεις το λόγο. Απλώς θα ήθελα να σας πω κύριε Πρόεδρε ότι εφόσον ψηφίσαμε ε, το εναλλακτικό κείμενο του ΕΛΚ στο πρώτο τμήμα της παραγράφου 41 πρέπει να διορθώσουμε τους καταλόγους του ε, ψηφοφορίας διότι το νέο παράγραφος 41 νέων καταπίπτει διότι είναι ακριβώς το ίδιο κείμενο. η επόμενη συμβιβαστική δηλαδή, στη σελίδα 5. Αναφέρεσαι στο 41α ή στο 41 σκέτο. Η συμβιβαστική 41α νέο καταπίπτει. Κύριε Πρόεδρε, αυτό δεν μας εμποδίζει να ψηφίσουμε το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 41, αλλά μιλάμε για το πρώτο τώρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε λοιπόν τώρα το δεύτερο τμήμα της 41. Ακριβώς. Και εδώ έχουμε δύο καταβιέρεση ψήφους. Okay. Also, zweiter Teil. Λοιπόν, το δεύτερο μέρος ψηφίζουμε τώρα. Εντάξει. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο δεύτερο. Η λέξη mandatory. Ποιος είναι υπέρ του όρου mandatory. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Απερίφθη κατά πλειοψηφία. Ερχόμαστε τώρα στο τρίτο τμήμα uh, with tax ranges. Υπέρ, κατά. Αποχές. Απερίφθη. Και τώρα ερχόμαστε στο τέταρτο τμήμα, with substantive indicative tax, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, το 41 νέο καταπίπτει, ερχόμαστε στο 42 σε δύο μέρη πρώτο μέρος. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 κατά αποχές εγκρίνεται 43 β πρώτο τμήμα κατά αποχές Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Τώρα ερχόμαστε στην παράγραφο 44 ε, εδάφιο 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 44α νέο και 44β νέο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 48α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 50α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 51β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 μαζί με την 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ερχόμαστε τώρα στην 57 ε, σε διάφορα τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι όντως εγκρίθηκε αλλά θα ήθελα να το δούμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος, 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 59 σε δύο τμήματα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62α εδώ έχουμε στο διορθωτικό κείμενο, στο κοριγκέντου, μία νέα ε, πρόταση την οποία θα ψηφίσουμε καταρχήν. Σας έχει διανεμηθεί. Είναι στην τρίτη σελίδα ε, και θα ψηφιστεί πρώτα. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Οπότε έτσι καταπίπτουν οι άλλες εναλλακτικές ε, της ιδίας παραγράφου και ερχόμαστε τώρα σε το εκτιμώντας FB υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε όταν ε, νομίζω ότι υπερψηφίστηκε αλλά στο δούμε ηλεκτρονικά υπέρ, κλείνει η ψηφοφορία εγκρίθηκε 24 υπέρ 14 ε, κατά. Ε, το EB ε, νέων υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τρίτο μέρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα έχουμε, ερχόμαστε στο τμήμα το οποίο έφυξε προηγουμένως η Περβόνσο. Ε, εγώ νομίζω ότι δεν χρειάζεται να ψηφιστούν αυτά τα θέματα. Περβόνς έχει το λόγο. Ζητάω να μην ψηφίσουμε τις τροπολογίες 126, 127, 313, 421, και 14, διότι καλύπτονται οι τροπολογίες αυτές. Για παράδειγμα, η τροπολογία 126. Κοιτάξτε την τροπολογία 126 και τι λέει και η παράγραφος 29 δέλτα, την οποία μόλις συγκρίναμε. Καταλαβαίνω ότι οι βουλευτέ θέλουν να λένε δύο φορέ το ίδιο πράγμα για να είναι σίγουροι ότι θα σε ακουστούν, αλλά εδώ καλύπτεται. Και οι άλλε καλύπτονται. Δεν χρειάζεται να τι ψηφίσουμε. Πολύ ε, σύντομα ε, θα ήθελα να παρακαλέσω την ομάδα των συντονιστών σχετικά με το θέμα 127. Μπαλτσίτης είναι από ποια πολιτική ομάδα και ε, η κυρία Γκουλάρ για το 27 αλλά Μπαλτσίτης για το 126. Και το 127 εντάξει. 126 λοιπόν. Όλε. Ε, δεχόμαστε αυτό να μην ψηφιστεί εφόσον ε, ε, συμφωνείς. Ε, ο Μπλοκ βέβαια. Μαργάριο και Ότμαρ, το 16 συμφωνείτε να μην ψηφιστεί. το 313 με συγχωρείτε ε, Σέτζο Κοφεράτη 421 ε, συμφωνώ να μην ψηφιστεί οπότε παραμένει ο Πασκάλ ε, όλοι λένε να μην ψηφίσουμε, να μην ψηφίσουμε, αλλά τώρα θα ψηφίσουμε για τα υπόλοιπα όλα μαζί. 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 ε, υπέρ κατά αποχές, αποχές ε, απερίφθη να ψηφιστούν όλα μαζί 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 124 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Όχι, δεν συμφωνούν να ψηφιστούν όλα μαζί. Λοιπόν, 133 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 252 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 275 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 300 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 367 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 382 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 395 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 396 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 397 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 398 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 403 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 406 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 456 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, ε, Εκτιμώντας 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 9 ε, ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 15 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 25 στο τέλος, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ε, και τώρα ψηφίζουμε ολόκληρη την έκθεση ηλεκτρονικά. Και είναι ε, δυνατόν ε, να ψηφίσουν όλοι. Ολοκληρώσατε. 31 υπέρ, 9 κατά, 2 αποχές. Συγχαίρουμε την Περβός. Χάνε Σόμποντα μου ζητά το λόγο. Έχουμε επιπλέον... Α, ναι, ναι. Ε, έχουμε περισσότερες υπέρ. Ε, συγχαίρω την Περβόσο διότι είχε μια ευρία πλειοψηφία. Όλα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά πραγματικά και στηρίξαμε τελικά την έκθεση. Πρέπει όμως να παραδεχτώ για την παράγραφο 57. Δεν ε, μας διευκολύνει τη ζωή. Πιστεύω ότι δεν είναι καλό να συζητάμε σήμερα κάτι τέτοιο στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ψηφίσαμε, αλλά να ξέρετε ότι θα τεθεί υποσυζήτηση στην Ολομέλεια δίχως άλλο. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Κάρας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους αυτούς οι οποίοι επί 1,5 χρόνια κατάφεραν να οδηγήσουν σε αυτή τη συνένεση, διότι η συνένεση ήταν η προϋπόθεση ε, για να θεωρήσουμε ότι καλύψαμε τις υποχρεώσεις μας. Και αυτό δεν, δεν αναφέρεται στο τι γίνεται σήμερα αλλά διότι ορισμένες από αυτές τις προτάσεις ίσως δεν υλοποιηθούν άμεσα αλλά πρέπει να ξεκινήσουν μεταξύ αυτών που το οποίο μπορούμε να πούμε σήμερα και τι χρειαζόμαστε στο μέλλον υπάρχουν δύο διαφορετικά θέματα και όσον αφορά τον προπολογισμό θα ήθελα να σας πω ότι στην Επιτροπή Σουρέ είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε επαρκή ε, χρηματοδότηση και τώρα αναφέραμε ένα αριθμό ο οποίος συνάδει με την Πολιτική Ένωση και με την Νομισματική Ένωση. Είναι όμως ε, μία από τις υποχρεώσεις μας προς ε, τους πολίτες να ολοκληρώσουμε την επιχειρηματολογία και να προχωρήσουμε εις ε, την ολοκλήρωση της χρηματικής και Χρηματοοικονομικής Ένωσης διότι έχουν εκφραστεί διάφορες απόψεις αλλά αυτό που είναι σημαντικό είναι να δείξουμε ότι το μέλλον της Ευρώπης δεν αναλώνεται σε καθημερινούς καυγάδες αλλά από κοινού είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε το έργο μας και την ένωσή μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα, λέει ο κ. Σκοφεράτη, να ευχαριστήσω την Περφόνς για την τεράστια προσπάθεια που έκανε, να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους συντονιστές. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα στο οποίο πλησιάζουμε έχει πολύ μεγάλο βάρος. Κάνατε κι εσείς μεγάλη προσπάθεια, Πρόεδρε, με τους συνεργάτες μας και έτσι φτάσαμε εκεί. Θέλω να υπογραμμίσω πάντως καταρχάς την συνέχεια στις προσπάθειες, στις προτάσεις και στις σκέψεις που κάναμε ανάμεσα στην ενδιάμεση έκθεση και σε αυτή την καταληκτική έκθεση. Υπήρξε μια φυσιολογική ανάπτυξη εξέλιξη της λογικής την οποία ξεκινήσαμε από κοινού εδώ και ένα χρόνο και. Και έτσι καταλήγουμε σε μια τελική πρόταση η οποία εγώ προσωπικά πιστεύω ότι θα είναι πραγματικά χρήσιμη σε όλες τις αρμόδιες επί της ουσίας επιτροπές που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το θέμα και να κάνουν προτάσεις δεσμευτικές για τις, επί των δικών μας προτάσεων. Εκεί όπου υπήρξαν ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες σε σχέση με ε, τις τροπολογίες που είχαν κατατεθεί, είναι προφανές εκφύσεως ότι ο καθένας από εμά αναγκάζεται θα έλεγα να εγκαταλείψει ένα τμήμα της αρχικής του έμπνευση και να δεχθεί μια νέα διατύπωση η οποία θα έλεγα εκφράζει με τον καλύτερο δυνατό σύνθετο βέβαια πάντα τρόπο την προσπάθεια η οποία έγινε. Ο συμβιβασμός λοιπόν στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι κάτι το αρνητικό. Δεν είναι αρνητικό εφόσον είμαστε σε θέση από κοινού να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάναμε έχει μια κάποια σημασία δίνουμε την ευκαιρία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές να ενισχύσουν και να ισχυροποιήσουν τα κριτήρια τα οποία ενέπνευσαν την έκθεση της Περβάνς. Το σημείο στο οποίο φτάσαμε είναι ένα σημείο το οποίο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί αντικατοπτρίζει την προσπάθεια την αποφασιστική που έκαναν όλοι και αντιπροσωπεύει και τις διαφορετικές τελικά πολιτικές ευαισθησίες, κάτι το οποίο είναι δύσκολο. Äh, Ευχαριστώ τον κύριο Κοφεράτη. Τελειώνοντας όμως θέλω να κάνω ένα σύντομο σχόλιο και μία, να εκφράσω μία ευχή και με αυτήν θα ξεκινήσω. Σε διάφορες συζητήσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια και με εκπροσώπους των κρατών μερών συναισθανθήκαμε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει μία πολύ κριτική τοποθέτηση σε σχέση με την Ευρώπη η οποία αυξάνεται αλλά υπάρχει και η επιθυμία να τελεσφορήσει ο στόχος της Ευρώπης και ελπίζω όλοι αυτοί οι οποίοι εδώ συμμετείχαν στην Επιτροπή βάσει αυτής της εκθέσεως ε, να μπορέσουν να δώσουν ένα μήνυμα εις τους πολίτες στις χώρες τους και να συζητήσουν ε, κατά τρόπον ώστε να συμβάλλουν ε, στο, ώστε να πιστούν και οι εθνικοί εκπρόσωποι, οι εθνικοί βουλευτές ε, για το στόχο μας διότι πολλοί δεν έχουν τους ίδιους, ε, τις ίδιες αξίες και τους ίδιους στόχους και μάλιστα αυτή τη στιγμή που πολλοί θεωρούν ότι η Ευρώπη δεν θέλω να πω ότι έχει αποτύχει αλλά ότι έχει φτάσει σε ένα διέξοδο πρέπει να είμαστε θαραλέοι και χωρίς καθυστέρηση να αποδείξουμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη ο Hans Dietrich Genscher που θα θυμάστε οι περισσότεροι από εσά και ο οποίος ε, έκανε μεγάλες προσπάθειες υπέρ του ευρώ πριν από δύο ή τρεις εβδομάδες έγραψε ένα άρθρο όπου είχε σαν επικεφαλίδα χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Και αυτό είναι και μας το σύνθημά μας. Αυτό που είπε ο Hans Ντίτριχ Genscher στην εφημερίδα Berliner Tagesspiegel πριν από δύο-τρεις εβδομάδες ουσιαστικά έλεγε ακριβώς αυτά τα οποία και εμείς πιο λεπτομερώς λέμε με την έκθεσή μας. Άρα Εάν κάποιος μας λέει ότι είσαστε τρελοί, ζητάτε πολλά ή παραφέρεστε, δεν είμαστε με νομοθετική επιτροπή και ως εκ τούτου δεν είναι κάτι το οποίο ζητάμε και σε μία εβδομάδα θα εφαρμοστεί ε, σαν νομοθεσία. Γι' αυτό διατυπώσαμε ελπίζω τολμηρές δηλώσεις. Ευχαριστώ όλους. Μία συμβιβαστική λύση είναι πάντοτε ένα συμβιβασμός κανείς δεν είναι 100% ευχαριστημένος, αλλά όλοι αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται κατά κάποιον τρόπο. Και τώρα έρχεται η φωτογραφία. Kollegen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Περβόνς βέβαια έχει το δικαίωμα και αυτή να πει ε, μια τελευταία λέξη. Άρα Περβόνς εσύ θα κλείσεις τη συζήτηση. Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι πόσο μεγάλη σημασία έχει τώρα που φτάνουμε στο τέλος της διαδικασίας αυτής η δουλειά που προσέφεραν όλοι, όλες οι πολιτικές ομάδες. Ως εισηγήτρια, λοιπόν, θέλω και εκ μέρους μου προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλους την Κοκομπού, κύριε Πρόεδρε, το σύνολο των συντονιστών, των σκιωδών εισηγητών, για όλο αυτό το χρόνο που συνεργαστήκαμε. Ξεκινήσαμε τις εργασίες μας και τότε κανείς δεν είχε αντιληφθεί το εύρος της κρίσης μέσα στην οποία βρισκόμαστε. Και με εκπλήσει που βλέπω ότι στο τελευταίο αυτό τμήμα της εργασίας μας όλοι κατάλαβαν, αισθάνθηκαν πόσο σημαντικό βάρος έχει το πολιτικό σκέλος και ότι εμείς οι ευρωβουλευτές θα πρέπει να κινητοποιηθούμε για να συνεχίσουμε το έργο αυτό που ξεκίνησαν οι ιδρυτές πατέρες. Ορισμένοι από εσά, δίχως άλλο, θα είδαν το web doc που έχει φτιαχτεί με τις εργασίες μας. Ε, στο τέλος έλεγε κάτι κάπως ρεαλιστικό αλλά και λίγο απογοητευτικό. Έλεγε οι προτάσεις της έκθεσης αυτής δεν θα γίνουν πραγματικότητα παρά μόνο εφόσον τις δεχτεί το Συμβούλιο και η Κομισιόν. Το ίδιο ισχύει και για αυτή την έκθεση. Αλλά Υπάρχει συνοχή με αυτό που ψηφίσαμε στην πρώτη έκθεση. Στην πρώτη έκθεση θέσαμε το πλαίσιο, το πνεύμα μέσα στο οποίο πρέπει να προσπαθήσει η Ευρώπη να βγει από την κρίση. Και σήμερα ε, καθορίζουμε τα μέσα για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς χωρίς να αλλάξουμε τίποτα από τη στρατηγική που εκπονήσαμε αρχικά και χωρίς να διστάζουμε για τα θέματα τα οποία είναι αρμοδιότητα άλλων επιτροπών. Πάντως, ημερίζουμε την πεποίθησή σας, Πρόεδρε, ότι σήμερα πρέπει να στραφούμε προς τους πολίτες ώστε οι προτάσεις αυτές να περάσουν στην πράξη και να αποφύγουμε τους ε, λαϊκισμούς οι οποίοι καραδοκούν. Σήμερα είμαστε στην υπηρεσία των πολιτών, των δικών τους επιθυμιών υπέρ μιας Ευρώπης η οποία να είναι στη δικιά τους υπηρεσία και όχι στην υπηρεσία μόνο των οικονομικών αγορών. Αυτό είναι και η βασική πρόταση της έκθεσης αυτής. Γιατί σήμερα, τρία χρόνια μετά την κρίση, πολύ συχνά οι πολίτες μας έχουν την αίσθηση ότι τελικά λίγα πράγματα έχουν αλλάξει και ότι αυτοί οι οποίοι διασώθηκαν στην αρχή είναι οι αγορές, οι οικονομικές αγορές και όχι οι ίδιοι πολίτες οι οποίοι βλέπουν σήμερα ότι ακριβένει η ενέργεια, ότι ακριβένουν λογαριασμοί που έχουν να πληρώσουν για τη θέρμανση, τις μεταφορές, οτιδήποτε και ότι δυστυχώς βρίσκονται και στην ανεργία. Αυτή είναι η βάση του μηνύματος που θέλουμε να στείλουμε βασιζόμενες στις προτάσεις αυτές. Ελπίζω να περάσει και στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή και ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε την ευκαιρία μετά από 1,5 χρόνο να ολοκληρώσω τις εργασίες αυτές. Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, μου είπαν ότι ο φωτογράφος έφυγε γιατί είχε ένα άλλο ραντεβού και καθυστερήσαμε. Θα βρούμε όμως φαντάζομαι έναν φωτογράφο και στο Στρασβούργο, οπότε... Α, λάθος, λάθος. Επανέρχεται. Θα περιμένετε άλλα πέντε λεπτά. Επανέρχεται. Λοιπόν, ε, πάρτε θέση.